15 και της κυρίας ήταν από 8 Ιανουαρίου οι οποίες ε, αντικαθιστούν τις κυρίες Νάιτ Σότεμπρουκ και τον κύριο Λουίς Ιντε αντιστοίχως. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις ευρωεκλογέ και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού του Κοινοβουλίου καλωσορίζω τις ε, συναδέλφους οι οποίες ε,